συζήτηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ας περάσουμε λοιπόν στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ σε ό,τι αφορά... Συγγνώμη, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν ήσυχα για να προχωρήσουμε κι εμείς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την πρόληψη χρήση των ε, δημοσιονομικών συστημάτων για, την, ε, για το ξέπλυμα ε, χρήματος χρήματο για τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας. Παρακαλώ, θέλουν να αποχωρήσουν, να το πράξουν ήσυχα για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Η τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος υιοθετήθηκε το 2015. Η Επιτροπή από το 2016 ζήτησε τα κράτη-μέλη να επιταχύνει την υλοποίηση μέχρι τα έτου του 2016. Στην τροποποιητική απόφαση του Ιουλίου 2016, οι τροποποιήσει αφορούν ε, τα ζητήματα χρηματοδότησης θερμοκρατίας και της διαφάνειας. Οι συνεισηγητές ε, έχουν υποβάλει 49 τροπολογίες και έχουμε 467 τροπολογίες συνολικά. Καλωσορίζω τους αδέλφους από την Επιτροπή ΕΚΟΝ και πιο συγκεκριμένα τον ε, κύριο Γαλτιέρη. Θα θέλατε να πάρετε το λόγο? Αλλιώς να δώσουμε το λόγο στους ε, συνεισηγητές. Just that, uh, να πω μόνο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Να πω μόνο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Υπήρξε σημαντική προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση. Θα ξεκινήσουμε το σύμμετρο δυνατόν τους τριμερείς διαλόγους. Θα θέλατε να προεδρεύσετε του πρώτου μέρους. Κανένα πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Κάρινς, εισηγητής για την Επιτροπή Οίκων. Ευχαριστώ πολύ. 459 ε, ε, τροπολογίες είχαμε την αρχή έκθεση και σχεδόν άλλες 320 στη συνέχεια κατατέθηκαν. Υπάρχουν ε, που εργάστηκαν σκληρά για την τέταρτη εκδοχή του κειμένου. Ε, πιστεύω ότι γενικά υπάρχει ομοθυμία ε, και ομονοούν όλοι στο βασμό που θέλουν να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομοποίησης ε, παρανόμων εσόδων. Κυρίως για τα άρθρα 30 και 31 Μητρό επιχειρήσεων και κυρίως για τα καταπιστεύματα, trust funds, ε, την τελευταία φορά δεν καταφέραμε να συμπεριληφθούν. Ε, αυτό είναι το γενικό πνεύμα των τροπολογιών. Έχουμε ήδη συναντηθεί με τους ε, συντονιστές δύο φορές. Ε, την άλλη εβδομάδα επίσης έχουν προβλεφθεί συσκέψεις. Νομίζω ότι οδεύουμε ολοταχώς προς τη δημόσια πρόσβαση σε αυτά τα μητρώα. Πιστεύω ότι στον τριμερή, σε επίπεδο συμβουλίου, θα συζητηθεί έντονα το ζήτημα των trust funds. Γιατί τα κληρονομικά, παραδείγματος χάρη, ε, για χρησιμοποιούνται παραδοσιακά τα καταπιστεύματα και δεν αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων. Φερρυπίν. Ε, τα μητρώα θα πρέπει να παραμείνουν όμως αποτελεσματικά και όπου υπάρχει ροή χρημάτων θα πρέπει να υπάρχει και καταγραφή Δεν θέλουμε εφεδρικά ε, συστήματα. Ίσως κάποιοι που συνέταξαν και κατέστησαν ανθρωπολογίες να διαφωνούν μαζί μου. Εγώ αυτό πιστεύω. Για τα άρθρα 30 και 31 θα μας απασχολήσουν πολλές τροπολογίες. Δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με τις συμβαστικές λύσεις, σίγουρα. Αλλά πάντως γενικά υπάρχει συμφωνία Επίσης πιστεύω δεν πρέπει περίτα να παρεμποδίζουμε ε, θεμητές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη με τις νέες διατάξεις και νομίζω ο συνεισηγητής θα συμφωνήσει. Δεν θέλουμε φυσικά τα ε, θεμητά συμφέροντα να τα παρεμποδίσουμε Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να βρούμε τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αναχέτηση παρανόμων δραστηριοτήτων, χωρί όμω να παρεμποδίζουμε και να παρακολύουμε την ε, φυσιολογική επιχειρηματική δραστηριότητα. Θέλουμε όλοι να ακολουθούν στου ίδιου κανόνε απλώ. Αν οι επιχειρήσει πρέπει να είναι σε μήτρο, ε, τότε και άλλε ε, αλλοδαπέ οντότητε ε, που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίση πρέπει να ακολουθούν στου ίδιου κανόνε κατευθυντήρε γραμμέ και να καταχωρίζονται στα μητρώα. Έχουν ε, καταδεχθεί πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Κάποιες δεν την προς την ε, απρόσκοπτη δημόσια πρόσβαση στα Μητρώα. μην ξεχνάμε ότι αυτή τη φορά το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε πώς θα καταφέρουμε να βρούμε αυτή την ισορροπία και κυρίως όταν αρχίσει ο τριμερής μετά το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη σίγουρα έχουν κάτι συμφέρον να προχωρήσει αυτή η νομοθεσία. Είναι ένα θέμα που πραγματικά αγγίζει την καθημερινή μας ζωή. Η Τζούδη Σαζεντίνη, λέει ο κύριος ε, Γκουαλτιάρη, είναι η συγγήτριά μας από τη Λίμπε. Ευχαριστώ πολύ. Για να προσθέσω κάποια πράγματα σε αυτά που είπε ο συνεισηγητή μου, ο Σέρφο Κάρεντσε, από τα εξή. Είσαστε παρόν όταν διαπραγματευτήκαμε την τελευταία φορά. Και καταφέραμε αυτό το αρχαίο να μπει, αρχαίο να μπει ε, στον ε, νόμο και είναι πολύ θετικό που τώρα η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει παραπέρα. Το Κοινοβούλιο με σωστή πλειοψηφία για μια ακόμα φορά θα συμφωνήσει ε, σε αυτή την κίνηση και επίσης θα συμφωνήσει με δημόσια μητρώα για τα καταπιστεύματα. Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όλες οι δομές οι οποίες λειτουργούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χώρες καταπιστεύματα. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι δομές οι οποίες λειτουργούν καλά ε, και με ποιο τρόπο. Αυτά είναι τα καλά νέα. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε έχοντας ε, στις συναντήσεις των οι σκιωδών επίσης θα συζητήσουμε και το θέμα των προπληρωμένων καρτών για επιγραμμικές και μη πληρωμές, online-offline. Και ε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα τρόπο με τον οποίο ταυτοχρόνως θα προστατεύουμε και τους πολίτες ε, αποκλείοντας όμως ταυτόχρονα ε, και τους τρομοκράτες από τέτοιες ε, δυνατότητες πληρωμής. Εγώ προσωπικώς ιδιαίτερος εκτιμώ όλες τις προσπάθειες αλλά θα πρέπει να είμαστε και σαφείς οι συνεισηγητές θα πρέπει να προωθήσουν έναν συμβιβασμό τέτοιο που να μπορεί να προσυπογραφεί από όλους ε, και να ακολουθήσει και το Συμβούλιο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς τη διαφάνεια ίσως να μην είναι αυτό που αποζητά το Συμβούλιο. Φαίνεται ότι τώρα ε, τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά ε, και ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει λόγω και των προσφάτων τρομοκρατικών συμβάντων ε, και των αποκαλύψεων για τα Panama Papers. Ε, ο κ. Γκουαλτιέρη, πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινέ θέσει, οι οποίε από ό,τι φαίνεται θα τύχουν μεγάλη συμφωνία. Ο κ. Ζήμων από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους εισηγητές. Είναι εξαιρετική η δουλειά που έκαναν και αποτελεί και πάρα πολύ καλή βάση για να βρει μια κοινή συμβαστική λύση. Είμαι αισιόδοξο. επόμενε συσκέψει των συντονιστών ε, θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε αυτή τη βάση και το χρειαζόμαστε κατεπηγόντω ε, μετά από τι αποκαλύψει ε, Παναμά. Ε, για τους σοσιαλιστές για αυτό το σχέδιο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Ε, χαιρετίζουμε καταρχάς το Μητρό ε, και ε, Φυσικά θα πρέπει να καταγράφονται όλοι οι οικονομικοί φορείς, όμως θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από τους συνεισηγητές, διότι κάνετε αυτή τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις συνήθεις επιχειρήσεις και τις παθητικές νομικές οντότητες. Εμείς θέλουμε να τοποθετήσουμε το όριο στο 10% του εταιρικού κεφαλίου και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο νόμονας για τα οικονομικά συμφέροντα των οντοτήτων. Ε, και Εκεί θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση και όλα αυτά θα πρέπει, όλες αυτές οι οντότητες θα πρέπει να ε, καταχωρίζονται στα μητρώα. Ε, και πέρα όμως από τους κανόνες θα πρέπει να προβλέψουμε και τις κυρώσεις. Για, για την πρόσβαση τώρα στα μητρώα, ε, για τις ε, επιχειρήσεις θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό που είναι διασυνδεδεμένα τα Μητρώα και υπάρχει πρόσβαση, αυξημένη μάλιστα πρόσβαση για τις επιχειρήσεις ε, και σίγουρα δεν γνωρίζει η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εθνικά σύνορα. Όμως προσοχή, θα πρέπει όλες οι αρμόδιες αρχές, οι υπηρεσίες, οι πληροφοριών και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα Μητρό για να μπορούν να κάνουν και εκείνη τη δουλειά τους. Ε, καταθέσαμε σχετικές τροπολογίες. Για όλες τις υπόλοιπες ε, νομίζω ότι, νομίζουμε ότι το μοναδικό κόλλημα ε, για αυτά τα Μητρώα είναι ε, το τέλος και η πρώτερη εγγραφή, διότι ε, δεν θέλουμε να υπερθεματίζουμε και να υπερβάλλουμε με το γραφειοκρατικό κόστος. Για το θέμα τώρα των trust funds, για να σχολιάσω και τη γραμμή των συνεισηγητών, θεωρώ επειδή πρόκειται για το πεδίο εφαρμογής και μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ήδη από τώρα μπορούμε να ε, στηρίξουμε την συμπερίληψη των ε, καταπιστευμάτων, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και πρόσβαση όλων, των, ε, όλων στο, στο, Μητρό στην τροπολογία 33 του εισηγήτη μιλάμε για μέτρα για τα κίνητα, για το ξέπημα βρώμικου χρήματος και για τέτοιες υπόγειες ε, δραστηριότητες. Θα την υποστηρίξουμε. Ε, πρέπει να δούμε τι κτηματολόγια υπάρχουν και τι μητρώα για τα ακίνητα για να δούμε αν είναι εφικτό αυτό. Επίσης για τα εκτεθειμένα άτομα. Ε, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στους πολιτικούς. Κοιτάξτε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Τα σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια μας δείχνουν ε, ότι σίγουρα θα ήταν ε, σωστό να μην περιοριστούμε στους πολιτικούς, στα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου ε, από τον αθλητισμό, από τις επιχειρήσεις, ε, από τη θρησκεία, διότι... Ξαναλέω, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεώσεις για όλους και σχετικές κυρώσεις για την πράξη κατά εξουσιοδότηση και τον μαύρο κατάλογο για τη, τους φορολογικούς παραδείσους. Έχαμε είχαμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπε ναι, ναι, αυτός ο κατάλογος είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κατάλογο της FATF. Ε, θα... Πρέπει όμως να διευρύνουμε αυτόν τον κατάλογο γιατί νομίζω ότι θα συναντήσουμε και στο μέλλον πρόβλημα εάν δεν αλλάξει κάτι. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χολμάιερ θέλει το λόγο. Είσαστε σκιώδης από το ΕΛΚ. Καλά τα λέω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι τώρα ε, σχηματίζεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή ε, ε, συμφωνούμε όλοι ως επιτοπλίστων, θέλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Φυσικά απ' έξω φαίνεται πολύ καλό να μιλάμε για τον αθλητισμό και να συμπεριλάβουμε διάφορα εκτεθειμένα πρόσωπα. Όμως μην ξεχνάμε ε, ότι πρέπει να έχουμε σχέση και με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει διαφθορά και δωροδοκίες και δωροδοσίες και δωροληψίες. Απλώς ε, ε, απαγορεύεται σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν προβλέπεται στην νομοθεσία, οπότε θα πρέπει να διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται, διότι μιλάμε και για την πρόσβαση στα έγγραφα και μιλάμε για επίσημα ε, καθήκοντα, επίσημα αξιώματα. Ποτέ, ποτέ δεν επιτρέπεται η διαφθορά και η δωροδοκία. Είτε πρόκειται για έναν ε, παίκτη του, ξέρω εγώ, για ταινίστα, ποδοσφαιριστή ή οποιοδήποτε άλλον. Έτσι. Αυτά απαγορεύονται από την ε, νομοθεσία και δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, να τους αναφέρουμε όλους ε, μεμονωμένα στον κατάλογο. Ίσως μόνο σε περίπτωση που έχει κάποια διαφορετική έννοια σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία. Οπότε μην κοιτάμε τα πράγματα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, αλλά από το πρίσμα της ε, ε, κείμενης νομοθεσίας. Δηλαδή, νομικά τι είναι υποχρεωτικό για να μπορέσουμε να ε, δράσουμε, να ανακόψουμε αυτές τις χρηματοδοτικές αιρώσεις που χρησιμοποιούνται για ε, ε, έκνομους σκοπούς. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ λίγο και στο θέμα της ε, τρομοκρατίας. Ε, μην ξεχνάμε ότι και η τρομοκρατία αλλά και το οργανωμένο έγκλημα, οργανωμένη εγκληματικότητα είναι τομείς όπου όταν μιλάμε για ε, φορολογικούς παραδείσους ή για ιδιαίτερα περίπλοκες οντότητες όπου ξεπλένονται χρήματα και κρύβονται λογαριασμοί και κεφάλαια Λοιπόν, ε, δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο σε αυτά γιατί μιλάμε για πώληση πετρελαίου, πολιτιστικών αγαθών. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται ε, για παράνομους σκοπούς για την ε, στήριξη και χρηματοδότηση τρομοκρατικών και εγκληματικών οργανώσεων και όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί μιλάμε τώρα για ένα τζίρο δισεκατομμυρίων. Οπότε θα πρέπει με τη νέα νομοθεσία να καταπολεμήσουμε και αυτές τις περίπλοκες χρηματοπιστωτικές οντότητες γιατί τίθεται ε, εν κινδύνο η ζωή ανθρώπων. Ευχαριστούμε, Γκόμες. Ναι, εμείς υποβάλαμε τροπολογίζει να υπάρχει δημόσιο μητρό των ε, δικαιούχων ε, των εταιριών και των καταπιστευμάτων με έναν ελάχιστο αριθμό πληροφοριών που να είναι δημόσια προσβάσιμες. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα όσα ανέφεραν οι συνεισηγητές μας, ότι έχουμε βρισκόμαστε σε καλή τροχιά για να πετύχουμε ε, αυτή τη συμφωνία και σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Επίσης, ε, καταθέσαμε τροπολογία, εγώ προσωπικά δηλαδή, και επιμένω σε αυτή τη τροπολογία, για να επεκτείνουμε το επαιδεί του Μητρώου και για τις αλλοδαπές ε, ε, επιχειρηματικές οντότητες ε, που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες που ήδη απαιτούν κάποιες τυπικές διαδικασίες όπως η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και έναρξη ενό τραπεζικού λογαριασμού. Νομίζω ότι αυτό θα επιτρέψει και θα μα βοηθήσει ιδίω να, ιδιαίτερω να αποκτήσουμε περισσότερη διαφάνεια. Και είναι σημαντικό όχι μόνο για την καταπολέμηση τη διαφθορά και τη φοροαποφυγή και του ξεπλήματο χρήματο, αλλά και για να αποτρέψουμε ε, το οργανωμένο έγκλημα, το διεθνέ έγκλημα και την τρομοκρατία να αξιοποιούν αυτέ τι ε, διαδικασίε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν γίνεται έτσι. Γίνεται μέσω πλασματικών και αληθινών εταιριών που αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία, αγοράζουν ε, γη και ακίνητα στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα σύστημα για να ξεπλένουν χρήματα. Οπότε μπορούμε να έχουμε ένα επίπεδο πληροφοριών για τα καταπιστεύματα, αλλά πρέπει να έχουμε και το ίδιο και για τις ε, εταιρείε ε, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ευρώπη. Και βασίζομαι και στο ΕΛΚ για τη στήριξή του. Ε, τροπολογίες άλλες αφορούν ε, πώς θα κλείσουμε ένα παραθυράκι στην ισχύουσα οδηγία, με την οποία ένας υψηλού επίπεδου μάνατζερ μπορεί να θεωρηθεί ε, δικαιούχος όταν δεν μπορεί να βρεθεί ο πραγματικός κάτοχος. Ρώτησα συναδέλφους πώς ισχύει αυτό. Είπαν ότι πρόκειται για σύσταση ενός φορέα. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αποδεκτό. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ήδη κατάχρηση και στη χώρα μου, πούμε, αυτό βλέπω. Το μοναδικό τμήμα τη ισχύουσης νομοθεσίας ε, που υλοποιήθηκε ή θεσπίστηκε μάλλον ε, από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2015 ήταν ακριβώς αυτό το παραθυράκι και δεν ήταν για καλό, σα διαβεβαιώ. Πρέπει να κλείσουμε λοιπόν αυτό το κενό και να μην ακολουθήσουμε τη σύσταση του FATCF ε, ως προς αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι οι οντότητε δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά με εντότητε των οποίων οι νόμιμοι κάτοχοι δεν είναι γνωστοί. Γιατί αυτό μα αποτρέπει από το να ε, αξιολογήσουμε αυτό το κίνδυνο. Το ίδιο ισχύει και για τα μητρώα των ιδιοκτητών, των νομίμων κατόχων. Δεν θα πρέπει να αποδέχονται την καταγραφή ε, εταιριών όπου μόνο ο senior manager ε, ταυτοποιείται. Από την άλλη, 10% των μετόχων θα είναι για μα μία ένδειξη νόμιμης κατοχής μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως ε, φύσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις οντότητες που θα πρέπει να ε, εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια, θέλουμε να διαβρύνουμε το πεδίο εφαρμογή και να ε, συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε παρέχει υπηρεσίες φορολογικής συμβουλευτικής ή ακόμα και νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ε, ε, έργων τέχνης κτλ ας μην γελιόμαστε. Αυτό ε, γίνεται όλο και περισσότερο ένας διαδεδομένος τρόπος ε, ε παράκαμψης ε, των ε, ελέγχων. Σε ό,τι αφορά τα εκτεθειμένα πρόσωπα, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε έναν επίσημο κατάλογο, το οποίο θα ετοιμάζεται και θα επικαιροποιείται από τα κρατημέλη και θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία από την Επιτροπή. Οι οντότητε αυτέ, τράπεζε κτλ., αυτή τη στιγμή αγοράζουν τι υπηρεσίε από αμερικανικέ ε, επιχειρήσει. Και πρέπει ε, να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή θα είναι αρκετά φιλόδοξη σε ό,τι αφορά την δικαιοδοσία και να μην ε, μεταγράψει απλώς τον κατάλογο FATF και έχουμε και τροπολογία, ούτω ώστε οι εθνικέ αρχές ε, να εφαρμόζουν μέτρα δέωσης επιμέλεια και για υπηκόου τρίτων χωρών που κάνουν αίτηση ε, υπηκότητα. Όπω είχαμε εδώ πριν για τη Μάλτα. Για προγράμματα IPP, χρυσέ θεωρήσει, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα ECR. Λούκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε η Σκιώδης από το ΕΛΚ, δεν πρόκειται για πραγματικά αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ε, είναι κοινό ο στόχο. Θέλουμε όλοι να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση τρομοκρατία, παράνομων δραστηριοτήτων, ε, ξέπημα βρώμικου χρήματο. Ναι, ε, πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μα και να άρουμε αυτό το πέπλο τη ανωνυμία, ούτω ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση από πλευρά του και να χρησιμοποιούν αυτέ τι χρηματοδοτικέ δράσει. Μέχρι αυτό το σημείο είναι πλήρη η ομοθυμία. Θα ήθελα όμω να σχολιάσω δύο ε, συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία ακόμη δεν υπάρχει ομοθυμία, τουλάχιστον με το ECR. Ε, πρώτο ζήτημα, η δημόσια πρόσβαση στα μητρώα αυτά ε, και οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, τους beneficial owners. Θα κατατέθηκαν πάρα πολλέ ε, τροπολογίε ασκήθηκε πίεση να είναι απολύτως ανοιχτή η πρόσβαση, δημόσια η πρόσβαση για όλους τους πολίτες, ε, αλλά νωρίτερα ε, οι ίδιοι, οι ίδιες προοδευτικές δυνάμεις χτυπιόντουσαν γιατί ήθελαν να προστατεύονται τα ατομικά δεδομένα και δεν ήθελαν λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Τα ξέχασαν όλα αυτά τώρα, οπότε ε, λέμε τώρα ότι ε, έχουν αξιώσεις και οι πολίτες και οι εμπλεκόμενοι ε, για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και τα καταπιστεύματα. Όταν μιλάμε για τα ονόματα ε, λοιπόν και για τις διευθύνσεις και για τα τηλέφωνα λέμε ότι πρέπει να είναι απολύτως δημόσια η πρόσβαση. Εγώ θεωρώ φυσικά ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για τις υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος και για όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για όλους όσους έχουν ένομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Αλλά μέχρι εκεί ε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σε αυτούς που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ένομο συμφέρον. Ε, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν. Δεν μπορούν να έχουν ένομο. Ε, συμφέρον. Παραδείγματο χάρη, ε, κάνουν, ε, προσπαθούν να βρουν πελάτε οι εταιρείε που προσφέρουν οικονομικέ υπηρεσίε. Γιατί λοιπόν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία ή εγκληματίε που θέλουν να κάνουν εκβιασμό επί τη βάση αυτών των στοιχείων, εν πάση περιπτώσει θέλουν να εκβιάσουν, να πιέσουν του έχοντε. Όταν κάποιο μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει ε, θύμα, ε, να, γίνει θύμα εκβιασμού, ε, τότε ναι, να αποκτήσει πρόσβαση, αλλά... Ε, ε, αντιστρέφουμε το βάρος της απόδειξης και πρέπει δηλαδή ένας ευημερών να αποδείξει ότι ε, πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση στα στοιχεία του για να μην υποστεί εκβιασμό. Ε, η σκιώδηση συγκήτρια του ΕΛΚ είπε ότι κατά πάσα περίπτωση δεν θα περάσει ούτε καν αυτό το ζήτημα από το Συμβούλιο. Οπότε βλέπουμε τι κάνουμε. Δεύτερο προβληματικό ζήτημα ορισμός των trusts ε, και αντίστοιχων ε, οντοτήτων. Προς το παρόν δεν υπάρχει ορισμός. Ε, λέμε ότι η οδηγία σχετίζεται και καλύπτει και τα trusts χωρίς να το ορίζουμε όμως. Και όλα τα συναφή και όλες τις συναφείς οντότητες χωρίς να ορίζουμε όμως τι εστί trust. Ο συνάδελφο Σβέν Κίκολτε είπε εχθές ότι βάσει ε, ε, για του γερμανικού δικαίου δεν καλύπτονται μόνο ιδρύματα αλλά και ενώσεις, ε, σωματεία με οργανώσεις, ιδρύματα τα οποία δεν θέλουμε εμεί να καλύψουμε με αυτήν την νομοθετική πράξη. παραδείγματο χάρη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δυσκολεύουν το άνοιγμα ενό νέου λογαριασμού, παραδείγματο χάρη, γιατί ε, πρέπει να δημοσιευθούν τα στοιχεία σε ένα δημόσιο μητρό. Θα πρέπει λοιπόν μέσα αυτήν την οδηγία να ξεκαθαρίσουμε ποιον καλύπτει το πεδίο εφαρμογή και ποιον όχι. Αυτά. Ε, σταματώ εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Μακόβι. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντώ. Ε, ως εισηγήτρια του ε, ε, ECR για την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ, ε, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να διατηρηθούν ε, οι τροπολογίες ε, για την διαφάνεια, κυρίως αυτές οι τροπολογίες οι οποίες αναφέρουν την ίχνη λασιμότητα και παρακολούθηση των συναλλαγών, καθώς επίσης και την εξέβρεση του πραγματικού κατόχου και πραγματικού ιδιοκτήτου. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε ε, και ε, κανονικά αρχεία όσον αφορά τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Θα πρέπει να προβλεφθεί και ε, πραγματική προστασία για τους whistleblowers όσον αφορά τις προπληρωμένες ε, κάρτες, ε, η χρήση τους ε, μέσω ίντερνετ αποτελεί πραγματικά, πραγματική απειλή για μας. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει απλώς να προβλεφθούν ε, κάποιες διατάξεις για τους πραγματικούς πελάτες τραπεζών ή πραγματικούς πελάτες που χρησιμοποιούν τέτοιες προπληρωμένες κάρτες. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να δημιουργήσουμε και ένα κατάλογο ε, των ιδρυμάτων που έχουν ε, διωχθεί και καταδικαστεί για παράνομες πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα ΑΛΤΕ, ο συνάδελφος Στόβατς. Τόρβαλτς. Θα μιλήσω αγγλικά, γιατί τα θα μιλήσω σουηδικά μάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές. Ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκαναν. Repetitias martyrios tudorum, όπως λέγανε και οι Λατίνοι. Νομίζω ότι ε, όλα αυτά, αυτά ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μετά από επανειλημμένες προσπάθειες τελικά μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση όπου υπάρχει ε, σχετική ομοφωνία. Και είναι και εξαιρετικοί συνεισηγητές μας και ε, γι' αυτό και τα καταφέραμε. Γνωρίζουμε την κατάσταση όπως ήταν ε, στο παρελθόν. Ε, και μπορούσα, μπορέσαμε λοιπόν με τις νέες προτάσεις ε, για να καλύψουμε τις τρύπε, τα κενά στη νομοθεσία ε, για τα φίντε ε, για τα, αυτά τα trust funds που εξακολουθούν να υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και λειτουργούν ως βιτρίνες για περίπλοκες χρηματοπιστωτικές οντότητες. Ε, όσοι έχουν, ξέρουν τη σειρά The Wire ε, ξέρουν ε, τι μπορεί κάποιος να κάνει με την ανωνυμία, με ανώνυμες ε, SIM κάρτες, ε, ανώνυμα, ανώνυμους λογαριασμούς. Είδαμε και το σκάνδαλο Παναμά που μας έχει οδηγήσει. Έχουμε και αυτό το πολύ beneficial owner ο πραγματικός ε, δικαιούχος ε, και παλέψαμε για να καλύπτονται και να συμπεριλαμβάνονται στα Μητρό και φαίνεται τώρα θα λειτουργήσουν εύρυθμα αυτά τα Μητρό και πίσω θα είναι δημόσια η πρόσβαση. Όμως ε, δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα έγγραφα Παναμά ξέρουν ότι μπορούμε να έχουμε σε ε, ε, ιδιοκτήτες ε, τέτοιων οργανισμών οντοτήτων που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ε, και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι ε, βούληση να κάνουμε κάτι για να καταπολεμήσουμε αυτές τις στάσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τις προσπάθειές μας και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε και πάλι ε, καλά αποτελέσματα για τα υπολοιπόμενα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ και τους συνεισηγητές κλείοντες. Σας ευχαριστούμε. Φάβιο Ντεμάζο για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εγώ αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στον πολιτικό και τον ποδοσφαιριστή, να σας πω ότι είμαι πολιτικός αλλά παίζω και ποδόσφαιρο, τα ξεκαθάρισα λοιπόν και τώρα ξέρετε πώς έχει η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ τους συνεισηγητές, φτάσαμε σε καλό συμβιβασμό και τουλάχιστον έχουμε συμφωνήσει και περί τίνος πρόκειται ε, να υπογραμμίσω ότι εδώ δεν πρόκειται να ε, πάρουμε θέση υπέρ ή κατά της επιχειρηματικότητας. Εδώ μιλάμε για τελείως άλλα πράγματα είδαμε και από την Europol στην Επιτροπή για τα Panama Papers ότι το μεγαλύτερο μέρος των ε, συνδιαλλαγών ε, ε, στα Panama Papers και σε αυτά που είχαν καταγεγραμμένα στα αρχεία τους είχαν κάποια σχέση με την τρομοκρατία. Επομένως μπορεί κανείς να πει ακόμα και στρεφόμενος προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι κάναμε ότι μπορούμε μπορούσαμε. Θα συμφωνήσω, όπω έχω συμφωνήσει και με άλλου στην Επιτροπή Panama Papers, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να βρεθούμε στη δύσκολη θέση να ξανακάνουμε τέτοια επιτροπή στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά το ε, θέμα που μα απασχολεί. Ε, πολλοί από του εμπειρογνώμονε στην Επιτροπή ε, Panama Papers, από τον Ζώζεφ Στίγκλιτς μέχρι, ε, μέχρι υπεύθυνου του FBI και της Europol, έχουν αναφερθεί στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος μία εταιρεία να μην θέλει ή να μην είναι σε θέση να πει ε, ποιο είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Και αν δεν μας πούν ποιος είναι ο κανονικό πραγματικό δικαιούχος, απλά να μην μπορούν να ε, ε, εμπορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξει και νομοθεσία που να ενσωματώνει και τι οντότητε που δεν είναι παρούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τώρα τα κατόφλια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε και εδώ πιο φιλόδοξοι γιατί ε, διαφορετικά μπορεί κανείς να διαλέξει τρεις-τέσσερις ε, ε, φίλους ή κάποια βολική νομοθεσία και μάλιστα ο κύριος Τίγλιτς πολύ καθαρά τα είπε όταν ήρθε στην Επιτροπή μας. Να υπογραμμίσω επίσης ότι θεωρώ ότι τις τελευταίες μέρες κάναμε μεγάλη πρόοδο. το θέμα, ας πούμε, του Freeport έχει καλυφθεί. Πιστεύω ότι οι εξαιρέσει ε, οι οποίες ε, ε, προβλέπονται στην νομοθεσία είναι πολύ σημαντικό που μπορούν τελικά να κριθούν ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτό είναι πολύ καλό. Και τέλος είναι πολύ θετικό που ε, αντιμετωπίζουμε και το θέμα του real estate, των περιουσιακών ε, ε, στοιχείων και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση των κτηματολογίων και των, των αρχείων real estate. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσει η Ολομέλεια ε, σχετικά με την απόρριψη του ε, καταλόγου. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες, ε, συγγνώμη, κάποιοι, κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους αυτούς που ξέρω ότι δουλεύουν πάρα πολύ σοβαρά και που τους ξέρω πολύ καλά γιατί έχουμε δουλέψει μαζί, να τους πω λοιπόν ότι αυτή η απόφαση που πήρε η ΕΚΟΝ και η ΛΥΜΠΕ να απορρίψει το τον ε, κατάλογο ε, αυτό ε, γιατί δεν έχουν ας πούμε συμπεριληφθεί χώρες όπως οι Μπαχάμες είναι μια σωστή απόφαση. Ε, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η νομοθεσία δεν είναι ε, πάντα ο σωστός. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε σε μια τέτοια λίστα να μην βρίσκονται χώρες όπως ε, ο Παναμάς ή η Μπαχάμες. Ευχαριστώ. from other groups, nor... Δεν βλέπω, λέει ο Πρόεδρος, να υπάρχουν αιτήματα αγόρευσης από, άλλες, από άλλους συναδέλφους. Επομένως δίνω το λόγο στον πρώτο εισηγητή. Ο κύριος Κάρινς. Ναι, θα ήθελα απλώς να πω πόσο εκτίμησα και ε, πραγματικά χάρηκα για τη συνεργασία με τους ε, συναδέλφους, ε, παρότι ήμασταν τόσοι πολλοί ε, στην κάθε συνεδρίαση. Ήταν πολύ παραγωγική, ενδιαφέρουσα και στοχευμένη συζήτηση που δεν συμβαίνει πάντα. Ιδίω όταν είναι πολύ άρθμη η αντιπροσωπεία. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από πλευρά Κοινοβουλίου. Όπως πάντα θα υπάρξουν και μεμονωμένα ζητήματα διαφωνίας. Εκεί που συμφωνούμε όμως σίγουρα είναι ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια νομοθεσία κατά της χρηματοδότησης της δημοκρατίας. Και οι διαφορές απόψεων γενικά είναι λιγότερο σημαντικέ σε σχέση με τον βασικό μας στόχο που είναι κοινό. Εγώ νόμιζα ότι εκπρόσωπο τη Επιτροπή δεν θέλει να πάρει το λόγο, αλλά βεβαίω και να τη το δώσουμε αφού τον ζητάει. Απλώ αν μπορείτε να είστε σύντομοι. Και μετά θα περάσουμε στου ε, υπόλοιπου ε, συνεισηγητέ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα από την ε, ομάδα της Γενικής Διεύθυνσης ε, Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση ε, του ξεπλήματος του οικονομικού χρήματος. Είναι πολύ καλό το έργο που έχει να παρουσιάσει το Κοινοβούλιο προς αυτό και ευχαριστούμε τους συνεισηγητές για την επικασματική αυτή τους εργασία. Θα μπορούσα να σταθώ σε πολλά σημεία, να εξηγήσω το σκεπτικό για, τον, για την αναφορά του senior manager όπου πάντα σκοπός ε, είναι να έχουμε κάποιο άτομο τουλάχιστον. Όμως αυτά είναι λεπτομέρειες, μπορούμε να βρούμε μια λύση προς αυτό. Δύο λόγια μόνο, γιατί το άκουσα την τελευταία παρέμβαση τον κύριο Ντεμάζη για τον κατάλογο ε, των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. Κατανοούμε τα όσα λέτε και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη μιας ε, ε, μεθοδολογίας για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως αυτό είναι μια χρονοβόρος διαδικασία. Προς το παρόν θα πρέπει να ενεργήσουμε επικοδομητικά. Δεν είναι το σημερινό μας ζήτημα βέβαια, διακόπτει ο Πρόεδρος. Α, μάλιστα. Ήθελα μόνο να πω Διακόπτω πρόεδρος και πάλι θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια αυτό το ζήτημα. Ε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Γκόμες, Σίμονς ε, και λοιπά ότι ελπίζουμε να υπάρχει μια πολύ καλή και θετική ψήφος ε, που θα δείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με κάθε σεβασμό δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ο κατάλογος ε, ε, τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. Κατά τη γνώμη μα. Θα δούμε όμως τι θα γίνει αύριο. Εδώ έχουμε ζητήματα της Επιτροπής Οίκων και της ΛΥΜΠΕ. Εγώ όμω είμαι και μέλος της Επιτροπής ανάπτυξη. και εμένα με απασχολούν οι παράνομες ε, ροές από την Αφρική και από άλλες χώρες όπου δεν καταβάλλονται φόροι, μεγάλες πολυεθνικές προσπαθούν να βρουν τρόπο να αποφύγουν ε, τη φορολόγηση. Αυτό είναι το βασικό μου κίνητρο και για να το κάνω αυτό χρειάζομαι διαφάνεια. Αυτό είναι ο βασικός μου στόχος και συνεχίζω να προσπαθώ να τον πετύχω. Προτείνω στο ECR οι δύο συνεισηγητές ε, να δουν ποια είναι η θέση τους ε, ως προς τη διαφάνεια, όμως γενικά νομίζω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία ε, που επιθυμεί την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ακόμα μία συνεδρία στις Κιωδών. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν μέχρι τότε. Αν θέλουμε να τηρήσουμε την προθεσμία, ε, για να έχουμε την ψηφοφορία στις 25 Γενάρη, σιγά σιγά στενεύουν τα χρονικά όρια. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Στις 25 Γενάρη προβλέπεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας συνεδρίασης.